περηφάνεια και μόνο να φτιάξει μια εσωτερική αγορά χωρί φιλοδοξία και τελικά κερδίζουν οι κερδοσκόποι, οι οποίοι τελικά αντικαθιστούν του μισθωτού, οι οποίοι ε, αμείβονταν από άλλου του οποίου εκμεταλλεύονται. Και οι δικαιούχοι, το διαπιστώνουμε, είναι έτοιμοι στα πάντα για να ε, διονυστεί αυτό το σύστημα. Εάν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάξει ε, πρότυπο, τότε θα την ξεκάνουν οι λαοί. Το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας φαίνεται ότι δεν φτάνει. Είμαι σίγουρη ότι οι ευρωεκλογέ θα είναι με δεύτερη προειδοποίηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κόχ, για ένα λεπτό παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν θέλουμε να ερμηνεύουμε αυθαίρετα και να κάνουμε κατάχρηση του ιστορικού μας κανονισμού, τότε εγώ φοβάμαι ιδιαίτερα. Αλλά να περάσω στο θέμα. Πριν από μερικέ μέρες, πήγα σε ένα πάρκινγκ στον αυτοκινητόδρομο Α4 στη Γερμανία και μίλησα με οδηγούς από διάφορες χώρες και ιδιαίτερα ε, με ορισμένους από την Πολωνία και την Ρουμανία και μου είπαν τα ίδια, ταυτόσημα. Πρώτον, θεωρούν ότι τους εκμεταλλεύονται και για πολλά θέματα όπως για παράδειγμα τους μισθούς και πότε θα γυρίσουν ε, στην ε, εστία τους φοβούνται να ρωτήσουν τους εργοδότες τους γιατί φοβούνται ότι θα χάσουν τη θέση τους. Είναι απάνθρωπες οι συνθήκες εργασίας τους. Ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται με αυτές τις εταιρείες γραμματοκιβώτια και το παράνομο καμποτάζ που στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Και τέσσερα, θέλουν οι κανόνες να είναι μη γραφειοκρατικοί και ελέγξιμοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Μην κλείνετε τα μάτια σας στην πραγματικότητα, διότι οι οδηγοί στους δρόμους μας πραγματικά τους αξίζει να βρούμε οικονομικές λύσεις για τα προβλήματά τους. Ακούστε τη βάση. Η κυρία Ρέγνα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις άθλιες συνθήκες εργασίας των οδηγών. Περί αυτού πρόκειται. <clears throat> Και εγώ κύριε Κόχ συζητώ με οδηγούς φορτηγών στα πάρκινγκ, στα αυστριακά σύνορα και ακούω περίπου αυτά που ακούτε κι εσείς. Μέρες κάθονται στο τιμόνι 15 ώρες ε, χωρίς διακοπή. Ζουν στα πάρκινγκ και κοιμούνται και εργάζονται σε ένα κουβούκλιο που είναι πολύ μικρό. Και το βράδυ θα πρέπει να προσέξουν να μην τους κλέψουν και τα το εμπορεύματά τους. Και όλα αυτά για μισθούς πείνας. Αν τους ρωτήσω τι θέλουν, τότε μου λένε θέλουμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, αξιοπρεπείς μισθούς. Να βλέπουμε την οικογένειά μας τακτικά θα πρέπει να μην επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ας ψηφίσουμε από κοινού για δίκαιε, συνθήκες εργασίας στους δρόμους μας. Για αυστηρού ελέγχους των χρόνων εργασία, διαλυμάτων και ανάπαυση. Μόνο έτσι θα δείξουμε το σεβασμό μας για τη σκληρή εργασία των οδηγών μας. Ο κύριος Φαντάλεν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση, προκειμένου οι οδηγοί μας να οδηγούν και να εργάζονται κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, για μένα, ότι πρέπει να φροντίσουμε να προβλέψουμε ένα πακέτο για την ασφάλεια. Όμως, τελικά διαπιστώνουμε ότι ο αγώνας είναι συνθήκες εξισορροπημένες προς τα κάτω όμως να έχουν τον ίδιο μισθό όλοι για την ίδια δουλειά. Αυτό είναι που είχαμε πει. Τώρα λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, δεν χειριζόμαστε καλά αυτή την υπόθεση. Μεροληπτούμε και στην νομοθεσία. Νομίζω ότι υπάρχει ελάχιστη επιθεώρηση. Έχουμε ελάχιστα στοιχεία στη διάθεσή μας. Ε, θα έπρεπε να υπάρχουν έλεγχοι διασυνοριακά και σίγουρα να μην υπάρχουν διακρίσεις. Και τέλος, έχουμε πάρα πολλούς παίκτες εδώ πέρα και αμφίβολες ε, διαδικασίες. Ευχαριστούμε κυρία Μέσινερ. Ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, στην εσωτερική αγορά μεταφέρονται πολλά εμπορέματα κάθε μέρα και πολλά οδικός. Περί αυτού πρόκειται. Θέλουμε πρώτα απ' όλα οδική ασφάλεια για τους οδηγούς μας. Γι' αυτό πρέπει να τηρούνται οι χρόνοι οδήγηση και ανάπαυση και θέλουμε και σωστέ συνθήκε εργασία. Και όπω είπαμε, υπάρχουν πολλέ εταιρείε γραμματοκιβώτια που δεν τι τηρούν. Υπάρχουν εταιρείε που αντιμετωπίζουν σωστά του οδηγού, αλλά δεν είναι όλε. Γι' αυτό θέλουμε παντού στην Ευρώπη να υπάρχουν σωστέ συνθήκε εργασία για όλου. Περί αυτού πρόκειται. Παράλληλα, ε, έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις και διαφορετικές περιοχές στην Ευρώπη και δεν πληρώνονται παντού οι ίδιοι μισθοί. Αλλά θέλουμε, επειδή έχουμε έλλειψη οδηγών, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας. Και τέλος, αυτό που θεωρώ ότι είναι κρίμα, είναι ότι οι οδηγοί λεωφορείων ε, τους ξεχνάμε. Και για τα λεωφορεία και για τα πούλμαν χρειαζόμαστε άλλους κανόνες. Ε, γιατί δεν είναι το ίδιο να, οδηγεί, να μεταφέρει κανείς εμπορεύματα ή ε, επιβάτες. Πρέπει και για αυτούς να βρούμε μια λύση. Η κυρία Βιώ, ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, και εγώ έχω εξοργιστεί διότι παρεμπόδιση τις τελευταίες ώρες της συζήτησης ε, και δεν ήταν σωστή. Όπως και στους μήνες δεν ήταν σωστή συζήτηση. Δεν δεν υπήρξε σωστή προσέγγιση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρω... Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ευρωβουλευτών και Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε υποσχεθεί πολλά πράγματα και δεν έχουμε ανταποκριθεί. Υπάρχουν κενά και γι' αυτό υπάρχει πάρα πολύ οργή, πάρα πολύ οργή. Ε, πιστεύω ότι το μέλλον τριών εκατομμυρίων των εργαζομένων στον τομέα είναι επιτάπητο και χρειάζονται ε, λύσει. Πρέπει να πλαισιωθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ. Πρέπει να πάμε από την πρώτη μέρα στην απόσπαση, να σταματήσουν ε, σταματήσει η κατάσταση στους αυτοκινητόδρομους. Είδα του οδηγού τι γίνεται και τα συνδικάτα των οδηγών που ζητούν ένα πακέτο κινητικότητα. Γι' αυτό για εκείνου που γι' αυτό ψηφιστήκαν σε αυτή την θητεία. Σε αυτή τη θητεία θα πρέπει να ψηφίσουμε. Ίσως η συσχετισμό δυνάμων στην επόμενη θητεία να μην είναι θετικό. Θα πρέπει να γίνει εντελώ διαφανώ η ψηφοφορία και θα πρέπει να σταματήσουν τα διάφορα προβλήματα και τα κενά. Λοιπόν, και το κείμενο για το καμποτάζ θα πρέπει να εξεταστεί πρώτο, διότι αυτό το κείμενο ψηφίστηκε στην Επιτροπή. Και ζητώ δημοκρατία να εφαρμοστεί πλήρω. Ο κύριος Μαρινέσκου έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θέλω ευρωπαϊκή ρύθμιση για ένα μοναδικό λόγο για να ξεφύγουμε από την εθνική νομοθεσία στη Γαλλία και τη Γερμανία που προστατεύει η νομοθεσία αυτή μόνο το δικό του τομέα. Αλλά θα ήθελα αυτή η ευρωπαϊκή ρύθμιση, η νομοθεσία να είναι ακριβοδίκαιη, να είναι διαφανής προς όφελος όλων των κρατών μελών και όχι μόνο προς όφελος κάποιων ε, κρατών μελών. Η πρόταση που έχουμε μπροστά μας είναι μια απόπειρα προστατευτισμού και μόνο για κάποιες ευρωπαϊκές περιοχές. Περιοχές Ευρωπαϊκής Ενώσεως και καλό τους συναδέλφους να μην κρύβονται πίσω από κοινωνικά επιχειρήματα. Εγώ ίδιο θέλω καλέ συνθήκε εργασία, πολύ καλέ συνθήκε εργασία για όλου αυτού που κινούνται σε αυτόν τον τομέα, εργάζονται σε αυτόν τον τομέα. Και μπορούμε αυτό να το ρυθμίσουμε. Ταυτόχρονα όμω θα πρέπει να καταργήσουμε όλα, όλες τις πρακτικές που είναι αντίθετες προς τις συνθήκες. Ε, θα πρέπει να σεβαστούμε την ελεύθερη διακίνηση, την ελεύθερη κυκλοφορία, παροχή υπηρεσιών κλπ. Και θα καλούσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει την νομοθεσία και να θεσπίσει για να προτείνει μια καινούρια σωστή. Ευχαριστώ. Ο κύριο Κρίστενσεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Κούλανεν, κύριε Τελίτσκα, κύριε Ερτογ, οι τρει σα στάσατε σε συμβιβασμό. Καλή βάση για μα για να βρούμε μια λύση, να βρούμε ισορροπημένου κανόνε να έχουμε κάτι που θα είναι καλύτερο, καλύτερε συνθήκε εργασία για του εργαζομένου, για του οδηγού στην Ευρώπη και να έχουμε θεμητό ανταγωνισμό των επιχειρήσεων στον τομέα. Και αυτό θα μα βοηθούσε να βελτιώσουμε την οδική ασφάλεια. Γι' αυτό ελπίζω ότι η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου να υποστηρίξει το έξοχο έργο που έκαναν οι συνεισηγητέ επί των τριών συμβιβασμών που πρέπει να ψηφίσουμε εντό του πακέτου. Νομίζω ότι είναι προφανές, είναι προφανές ότι τώρα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε καταστροφικές δυνάμεις και κάνουν ό,τι μπορούν ούτω ώστε να μας εμποδίσουν από το να πετύχουμε μια λογική συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχουν εκείνοι που θέλουν να ανταγωνίζονται σε κακές συνθήκες που επιβάλλονται στους οδηγούς. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι στόχος μας. Μην το δεχτούμε αυτό και ας ψηφίσουμε τις συμβαστικές και έτσι θα καταλήξουμε σε μια λογική λύση. Ο κύριος Κιουτσούκ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι. Είναι καλό που διεξάγεται αυτή η συζήτηση, διότι αναδεικνύονται διάφορες απόψεις και πόσο περίπλοκο είναι το θέμα. Το πακέτο της κινητικότητας 1 αντιβαίνει της ιδέας της ενιαίας αγοράς. Αυτή η προσέγγιση στο πρόβλημα δεν οδηγεί στην ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς, αντιθέτως την υπονομεύει. Βεβαίως, αξίζει στους οδηγούς να έχουν καλές συνθήκες εργασίας. Είναι ένα υπεύθυνο επάγγελμα, δύσκολο επάγγελμα, αλλά δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό καταστρέφοντας επιχειρήσεις, ένα τομέα που αναπτύχθηκε βάσει των αρχών της ελεύθερης αγοράς και στη χώρα μου και μόνο αφορά το 17% του ΑΕΠ και, παρά, ε, και δίνει δουλειά σε 500.000 ανθρώπους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ισχυροποιηθεί ε, μέσω ανταγωνισμού κέντρου ε, κατά της περιφέρειας. Η απόρριψη δύο από τα τρία χαρτοφυλάκια δείχνει ότι υπάρχει έλλειψη συνένεση όσον αφορά το πακέτο υπό τη μορφή που έχει και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας ανευθυνότητα και να τα υιοθετήσουμε ανεύθυνα. Διότι αν κάνουμε κάτι τέτοιο θα έχει αρνητικότατο αντίκτυπο για εκατομμύρια ανθρώπου. Η κυρία Σμιτ έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και έτσι βλέπουμε ότι πολύ γρήγορα μπορεί το Κοινοβούλιο να μην είναι σε θέση να αποφασίσει αν ο καθένας ε, περιχαρακώνεται στους εθνικούς εγωισμούς του. Γιατί τότε μόνο ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής μας μένει. Πρέπει να επιδιώξουμε όμως ε, τις καλύτερες λύσεις, τις ευρύτερες και αυτές να αποφασίσουμε. Αυτό δεν το καταφέραμε στις πολιτικές ομάδες, οπότε και στις επιτροπές. Οπότε και εδώ στην Ολομέλεια αποτύχαμε. Ο ιστορικός κανονισμός ε, εφαρμόστηκε και τραβήχτηκε ούτω ώστε να γίνει αγνώριστος. Και βλέπουμε που καταλήξαμε και πόσο τοξική είναι η κατάσταση και πόσο ε, υπερασπίζει το καθένα στα δικά του συμφέροντα. Ε, εάν ε, ε, συνεχίζουν όλοι να βασίζονται μόνο στα δικά του συμφέροντα και κάθε διαφορετική αντίληψη να την θεωρούν εμπόδιο. Αυτό οδηγεί σε νέο προστατευτισμό. Και στην ομάδα μου και παντού έτσι θίγουμε την Ευρώπη. Δεν υπάρχουν συμβιβασμοί ε, στην Επιτροπή Τραν παρά μόνο για το καμποτάζ. Ε, κύριε, κύριε Μπρέσο, έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το πακέτο κινητικότητα είναι καρπό κοπιαστική εργασία που έγινε από τι αρμόδιε επιτροπέ για να θέσει κάποια τάξη σε ένα τομέα που χαρακτηρίζεται από άγριο ανταγωνισμό, που όχι μόνο δημιουργεί απαράδεκτε συνθήκε διαβίωση για του οδηγού, αλλά θέτει σε κίνδυνο επίση τη ζωή όλων των Ευρωπαίων πολιτών στου δρόμου και συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στι εκπομπέ του άνθρακο. Εν αναμονή τη διαθυμότητα σιδηροδρομικών μεταφορών, που θα είναι τομέα ισχυρό και θα είναι ταχύε οι μεταφορέ, χάρη στα διευρωπαϊκά δίκτυα και έτσι να μειώσουμε τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακο από του δρόμου μα, πιστεύω εν τω μεταξύ είναι απαραίτητο να καταλήξουμε σε λογική συμφωνία, να εξυγχρονίσουμε τον τομέα και να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την ποιότητα εργασία για του οδηγού Πιο συγκεκριμένα, η θέσπιση, η πολύ αρχική του εφιούς ταχυγράφου θα επιτρέψει διεξαγωγή αποτελεσματικών ελέγχων. Θα μπορούμε να εγγυηθούμε ότι γίνονται σεβαστές οι προδιαγραφές και οι κανόνες. Πιστεύω λοιπόν συνάδελφοι ότι θα πρέπει να έχουμε το θάρρο να ψηφίσουμε και να ε, δείξουμε κατά πόσο το Κοινοβούλιο σε τόσο σημαντικά θέματα είναι ικανό να λάβει μια απόφαση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Ντεγκράντε Πασκουάλ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ό,τι πετύχαμε στην Επιτροπή Μεταφορών ήταν μια ευαίσθητη ε, ισορροπία η οποία απορρίφθηκε τελικά. Κατά τη γνώμη μου, και το λέω με κάθε σεβασμό, έχει να κάνει με σαφή συμφέροντα κάποιων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βάζει εμπόδια στις πιο περιφερειακές ε, χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός. Τώρα, καταφέραμε τελικά να υποστηρίξουμε ένα dumping κοινωνικό με αυτές τις συμφωνίες. Αλλά είμαστε κατά της ελεύθερης αγοράς και υπάρχουν επιχειρήματα τα οποία τελικά κρύβονται γιατί ουσιαστικά πρόκειται για τα συμφέροντα των χωρών μελών κατά τον προστατευτισμό. Δεν προσφέρουμε πιο αξιοπρεπεί συνθήκες. Τόσα λέμε για την ανάπαυση στην καμπίνα των φορτηγών, τα περικαμποτάζ, οι διοικητικέ ε, διαδικασίες, ο χρόνος εργασίας, τα ελαφρά οχήματα και το πεδίο εφαρμογή της νομοθεσίας θα έχουν σαν αποτέλεσμα περισσότερο κόστος στις μεταφορές που θα κάνουν ε, οι επιχειρήσεις που δρούν στις περιφερειακές χώρες. Γι' αυτό διακόπτη πρόεδρος. Εύχομαι κάθε επιτυχία παρόλα αυτά. Ο κύριος Λιμπεράτσκι. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Εύχομαι να είχαμε άλλους τρεις τη Δευτέρα, ώστε να είχαμε απορρίψει οριστικά το κείμενο αυτό. Η γνώμη μου είναι ότι εδώ δεν πρόκειται πραγματικά για το χρόνο οδήγηση, την ανάπαυση, του οδηγού κτλ. Πρόκειται για να περιορίσουμε την πρόσβαση στην αγορά σε κάποιο τμήμα τη Ευρώπη ε, που αποδείχθηκε ότι ήταν αρκετά ανταγωνιστικό. Οπότε αυτό το οποίο μας λέτε τώρα είναι ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και αν είσαστε ανταγωνιστικοί τότε θα σας βάλουμε εμπόδια. Αν Ακούω τώρα ότι κάποιες χώρες ε, μέλη μονομερός θα δράσουν αν δεν περάσει τελικά αυτό το πακέτο, νομίζω ότι αυτό είναι καθαρά εκβιασμός. Αυτοί που λένε τέτοια πράγματα πρέπει να το ξέρουν ότι οι εργαζόμενοι τους οποίους υποστηρίζουν δεν είναι στην πραγματικότητα αποσπασμένοι. Ας αφήσουμε αυτό την προσπάθεια να την αφήσουμε για την επόμενη θητεία. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό κυρία Γιασλοβέσκα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εδώ συζητάμε κατά πόσο το πακέτο αυτοκινητικότητας μπορούμε να το ψηφίσουμε τώρα ή όχι. Αλλά έτσι κρύβουμε το θέμα του συντονισμού ε, συστημάτων ασφάλειας. Στο άρθρο 14 τα κριτήρια που περιλαμβάνονται ε, μιλάνε για την απόσπαση. Τελικά όμως οι διεθνείς επιχειρήσεις δεν μπορούν να τηρήσουν τα κριτήρια αυτά κάθε εργοδότης διακινδυνεύει με κάθε αλλαγή της νομοθεσίας αναδρομικά. Μία γαλλική επιχείρηση δηλαδή μπορεί να αναγκαστεί να ε, εργάζεται πάνω κάτω μάλλον από τις συνθήκε του της γερμανικής νομοθεσίας ή άλλης. Καταλαβαίνετε τι χάος θα δημιουργηθεί εφόσον εφαρμοστεί τελικά το πακέτο αυτό χωρίς το 14 πρέπει να το ξαναδούμε το πακέτο και να φροντίσουμε για αλλαγές που θα επιτρέπουν στις οδικές επιχειρήσεις να δρουν χωρίς εμπόδια στην εσωτερική αγορά. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε υπεύθυνοι για τις λύσεις εκείνες που θα διευκολύνουν τη ζωή μας μέσα στην εσωτερική αγορά με λιγότερο διοικητικό βάρος για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, κυρία Γιονγκέριους. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εδώ στο Στρασβούργο σήμερα στις Βρυξέλλες, στις άλλες διαδηλώνουν οι εργαζόμενοι γιατί θέλουν ένα αξιοπρεπές μέλλον. Και έξω από αυτή την αίθουσα να ξέρετε ότι κανένας δεν καταλαβαίνει τι προσπαθούμε εμείς να κάνουμε και χάνουμε έτσι την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στις Βρυξέλλες. Αλλά δεν πρόκειται μόνο γι' αυτό. Είτε σήμερα, είτε τον Απρίλιο, είτε αργότερα, δεν έχει σημασία πότε θα ψηφίσουμε, αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι να πληρώνονται αξιοπρεπώς οι εργαζόμενοι και να αναπαύονται όπως πρέπει. Οι οδηγοί των φορτηγών και των λεωφορείων τώρα μπαίνουν σε ανταγωνισμό μεταξύ τους. Ποιος θα ζητήσει το χαμηλότερο μισθό για να μπορέσει να δουλέψει. Δεν πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τους ε, οδηγούς, να σταματήσει αυτό και επίσης να σταματήσει και αυτή η ιστορία με τις επιχειρήσεις εικονικής έδρας. Γιατί μόνο τότε θα μπορέσουμε να προσφέρουμε αξιοπρεπείς συνθήκες στους εργαζόμενους μας. Ευχαριστούμε κυρία Μωρέ, σε ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, το έργο που κάνουμε και η συζήτηση που διεξάγεται σήμερα το πρωί αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Επίσης όμως αφορά, όσον αφορά αυτά που είναι εκτός του διεθνούς εμπορίου, αφορά και τις συνθήκες ε, που αφορούν τους αποσπασμένους εργαζομένους. Έχουμε μια οδηγία όσον αφορά, μια γενική οδηγία έχουμε πλαισίωσης ε, της αποσπασμένης εργασίας. Όμως με τους οδηγούς του μεταφορικού τομέα. Δεν μπορούμε να έχουμε αποσπασμένου εργαζομένου πρώτη ε, τάξη και δεύτερη τάξη, πρώτη κατηγορία και δεύτερη κατηγορία, όσον αφορά το μισθό και την κοινωνική προστασία. Είναι ο τομέα τη της κοινωνική Ευρώπη. Θα πρέπει τι διεθνεί μεταφορέ να τι ρυθμίσουμε, το καμποτάζ, να μην υπάρχει αναδίπλωση εθνική και αποφάσεις που μπορούν να διαλύσουν την Ευρώπη. Θα πρέπει να να φτάσει λοιπόν στο σωστό επίπεδο η νομοθεσία. Αυτή είναι η Ευρώπη των πολιτών, αυτή είναι η Ευρώπη των εργαζομένων, αυτή είναι η βάση της Ευρώπης πάνω στην οποία να εμείς πρέπει να κινηθούμε και να εργαστούμε. Ο κύριος Κουρουμπάσεφ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρόεδρο Ταγιάννη που έλαβε τη μόνη δυνατή απόφαση. Ούτε υποστηρίζει εκείνους που είναι υπέρ, ούτε εκείνους που είναι κατά του πακέτου. Ο πρόεδρος είναι απλώς υπέρ του νόμου. Αρκετές φορές εκβιαστήκαμε μέσω δηλώσεων που έλεγαν ότι αν δεν εγκριθεί το πακέτο, τα κράτη-μέλη θα λάβουν τις δικές τους αποφάσεις. Είναι Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή ή είναι Ένωση εθνικών κρατών που είναι συναθρισμένα σε διάφορες ομάδες. Ε, είδαμε το κοινωνικό dumping σαν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι δυτικές επιχειρήσεις άρχισαν να πληρώνουν μισθούς που είναι η μισή του κανονικού μισθού σε οδηγούς από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Για να αποφευθεί αυτή η μάχη και να μην συζητήσουμε το πακέτο και να μην το ψηφίσουμε τώρα, δεν δείχνει αδυναμία. Θα συνεχίσουμε τη μάχη για το πακέτο κατά τη διάρκεια αυτής αλλά και της επόμενης ε, θητείας. Μοντέιρο Ντε Αγιάρ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συζητούμε το πακέτο κινητικότητας. Προφανώς είναι πολιτικός πώς ακαθόδες θέμα αλλά έχει γίνει ολόκληρο μυθιστόρημα που κρατάει χρόνια. Πρέπει να σεβαστούμε το έργο των συναδέλφων στι διάφορε επιτροπέ και των εισηγητών, κυρίω το έργο τη Επιτροπή Μεταφορών. Η διαδικασία που ακολουθεί το Κοινοβούλιο τώρα δεν είναι δημοκρατική και δεν εναπόκειται σε εμά να αναλύσουμε 1.700 τροπολογίε που κατετέθησαν τελευταία στιγμή. Όταν αυτή η πρόταση έφτασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ήδη μεροληπτική αυτό σήμαινε ότι όλο το έργο που έγινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν μια προσπάθεια εξισορρόπησης του προϊόντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν ήταν ισορροπημένο και πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η ενιαία αγορά και ελεύθερη διακίνηση των αγαθών και των εργαζομένων Είναι ο στόχο να υπάρχει αυτή η ελεύθερη κίνηση. Καλύτερα να μην έχουμε συμφωνία παρά να έχουμε μια κακή συμφωνία. Και ελπίζω ότι η επόμενη θητεία θα καταλήξει σε καλύτερη συμφωνία που θα έχουμε μπροστά μα. Λοιπόν, θα παρακαλούσα σε αυτού που είναι στου διαδρόμου και που συζητούν, αν μπορούν να κάνουν ησυχία και να σταματήσουν συζητήσει, να τι κάνουν εκτό ημικυκλίου. Η κυρία Σαπαρτέλντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να έχετε επίγνωση του γεγονότο ότι το πακέτο κινητικότητα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά από του συναδέλφου ε, οι συγητέ θα σημάνει τη χρεοκοπία εκατοντάδων μεταφορικών επιχειρήσεων στην Ανατολική Ευρώπη και θα χαθούν πάρα πολλέ θέσει εργασία. Θα υπάρξουν συνέπειε όχι μόνο επί των μεταφορικών εταιριών τη Ανατολική Ευρώπη, θα υπάρξουν και αρνητικέ συνέπειε όσον αφορά τη λειτουργία τη ενιαία αγορά. Θα έχουν περισσότερο προστατευτισμό και στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό είναι απαράδεκτο, αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει κληρονομιά της 8ης θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, θα πρέπει να προστατεύσουμε όλοι τα κοινωνικά δικαιώματα των οδηγών του μεταφορικού τομέα. Αλλά οι συνάδελφοι που χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα θα πρέπει να συμφωνούν επίσης και μια τιμή ανά χιλιόμετρο που θα είναι δίκαιη. Ε, σωστή που θα επιτρέπει στις εταιρείε των περιφερειακών χωρών να καλύπτουν το κόστος και να εγγυώνται συνθήκες εργασίας που θα είναι καλύτερες. Πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι. Ε, δεν θα πρέπει να υπάρχουν πολύ αυστηροί όροι για την επιστροφή και για την απόσπαση. Συγχωρείτε σας ε, διακόπτω, λυπάμαι. Νόβακοφ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ορισμένοι στηρίζουν αυτό το πακέτο και ισχυρίζονται ότι αγωνίζονται για τους εργαζόμενους του κλάδου. Μα γιατί αγωνίζονται, με πώς αγωνίζονται. Στην ουσία θα καταστρέψουν τον τομέα αυτό. Ε, ελέγχθη ότι οι συμβιβασμοί που επετέφθησαν είναι μια σωστή βάση για να υπάρξει ψηφοφορία. Δεν ισχύει. Κοιτάξτε, δεν μπορεί ο, από μόνοι μα να αποφασίσουμε, γιατί δεν είναι παρόντε όλοι αυτοί που πρέπει να αποφασίσουν. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Κοινοβουλίου, ένα ε, εισηγητή αρνείται εντελώ την έκθεση που υποτίθεται ότι παρουσιάζει. Κοιτάξτε, Έχουμε τρει εβδομάδε μέχρι τη λήξη τη θητεία. Δεν υπάρχει χρόνο για να υπάρξει μια σωστή συζήτηση και σωστή λύση. Η μόνη δυνατότητα είναι να αναβληθεί για το επόμενο κοινοβούλιο που θα έχει πέντε χρόνια να το συζητήσει. Δεν είναι πια θέμα μεταφορών, αλλά κοινή λογική. Είναι η τέταρτη προσπάθεια που γίνεται να περάσει αυτό το πακέτο και θα αποτύχει και αυτή. Αυτό θα πρέπει να μα κάνει να καταλάβουμε περί τίνο πρόκειται και πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα. Πολλά επετέφθησαν, αλλά πάρα πολύ περισσότερα πήγαν στραβά. Α το αφήσουμε για την επόμενη θητεία. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους ε, τους συζητητές, αλλά να αναφέρω το εξής. Αποτύχαμε. Δεν καταλήξαμε σε συμβασμό. Δεν είναι συμβασμό αυτό που έχουμε μπροστά μας. Έχουμε 1600 τροπολογίες. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει συνένεση. Και λύγει και ο χρόνος. Δεν έχουμε χρόνο. Τι μας μένουν, τρεις εβδομάδες. Άρα τι λύση μπορούμε να βρούμε. Μια λύση που να βασίζεται στις εξής αρχές. Πρώτον, πρέπει να υπάρξει συμφωνία και επί των τριών εκθέσεων, γιατί αλληλοσυνδέονται. Εάν δεν συμφωνηθούν όλα, δεν μπορεί να έχει συμφωνηθεί τίποτα. Δεύτερον, πρέπει οι κανόνες ε, που θα αποφασίσουμε να ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους και όλους τους μεταφορείς για να λειτουργήσει σωστά η ενιαία αγορά. Και φυσικά πρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας των ε, οδηγών, την οδική ασφάλεια. Όλοι τα επιδιώκουμε αυτά. Αλλά δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε κάποια κράτη-μέλη και κάποιοι μεταφορείς να εξαιρούνται. Ο κύριος Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ. Είχα την ευκαιρία να εργαστώ ως υπουργό Μεταφορών και γνωρίζω πολύ καλά τον τομέα. Δεν θα προβώ σε δηλώσεις. Αναμφιβόλα θέλω να πω ότι οι κοινωνικές εγγυήσεις για τους εργαζομένους είναι υψής της σημασίας. Σωστά αναφέρθηκε ότι μια διχασμένη ενιαία αγορά σημαίνει ότι οι εταιρείε από τις περιφερειακές περιοχές δεν μπορούν να προσεγγίσουν τι μεγαλύτερε αγορέ. Αν λάβουμε αυτή την απόφαση και ευχαριστώ τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Ταγιάννη, που έλαβε σοφή απόφαση, που αποφάσισε να μην διεξαχθεί ψηφοφορία, λέω όμω ότι θα ήθελα να ενθαρρύνω να ενδιαφερθούμε για το εξή θέμα, ότι οδηγεί από την Λιθουανία, την Εστονία και μικρές, από μικρέ χώρε που εργάζονται σε επιχειρήσει μεγάλων εταιριών, όπω είναι μεγάλων χωρών, όπω είναι η Γερμανία και η Ολλανδία, πληρώνονται τον ίδιο μισθό όπω οι πολίτε αυτών των χωρών. Μπορούν να επιστρέψουν το Σαββατοκύριακο στο σπίτι του. Έχουν τη δυνατότητα να διαμένουν προ ανάπαυση στα ξενοδοχεία. Διακοπή. Πρέπει να ολοκληρώσετε. Ο κύριο Λίνκρεν. Και παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη να είσαστε ήσυχοι όσο μπορείτε. Αυτή η συζήτηση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. σα παρακαλώ. Κύριε Λίνκρεν, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι μια μεγάλη τραγωδία. Η οικονομία των μεταφορών στην Ευρώπη περιμένει από το Κοινοβούλιο να λάβει μια απόφαση στο συγκεκριμένο τομέα. Τι κάνουμε, τους παρατάμε, αφήνουμε τους εργαζομένους στη μοίρα τους, τους αφήνουμε για να στηρίξουμε το κεφάλαιο, περί αυτού πρόκειται. Πρόκειται περί του γεγονότος ότι πολλά πολλά μέλη του Κοινοβουλίου υπερψηφίζουν του να οδηγούνται τα φορτηγά από οδηγού άλλων χωρών. Εγώ είμαι Σουηδό. Δεν πιστεύω ότι είναι αποδεκτό εμεί να έχουμε 2.000, 3.000, 4.000 αλλοδαπά οχήματα στη χώρα μου, φορτηγά που είναι συνεχώ στου δρόμου και εκτελούν εσωτερικέ μεταφορέ. Αυτό είναι επιζήμιο για την αγορά, την ενιαία αγορά και την, εσω... και την τόπια αγορά. Και σίγουρα αυτό δεν θα πρέπει να είναι ο στόχο τη ευρωπαϊκή συνεργασία το γεγονός ότι όλες οι χώρες θα πληγούν από το ίδιο πρόβλημα που βλέπουμε τώρα. Πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Η κυρία Βόλτμανς έχει το λόγο. Κυρία Βόλτμανς, ζητήσατε το λόγο, όχι, ωραία. Ο κύριος Πιμέντα Λόπες έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο χαοτικός τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το πακέτο δείχνει σαφώς το πώς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στρεβλώνονται όποτε προσπαθούν να προστατεύσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Το να υποβληθούν αυτές οι προτάσεις και βλέποντας ταυτόχρονα και τις κατευθυντήριες γραμμές του ε, Συμβουλίου βλέπουμε ότι η ονή δεν είναι καλή. Το να χρησιμοποιούμε τα δικαιώματα των εργαζομένων σαν δικαιολογία για αυτή τη μορφή κανονισμού, αυτή τη μορφή νομοθεσίας περί καμποτάζ, και να αντιμετωπίζεται έτσι ο χρόνος ανάπαυσης και ο χρόνος εργασίας δεν είναι σωστός. Σημαίνει ότι μπορεί να παραταθεί από δύο σε τρεις ή τέσσερις εβδομάδες η περίοδος κατά την οποία οι οδηγοί θα πρέπει να οδηγούν χωρίς να αναπαύονται σωστά και να έχουμε ανάπαυση ενός Σαββατοκύριακου. Αυτό είναι μια άμεση επίθεση κατά των δικαιωμάτων των εργαζομένων κατά την απόψή μου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, κυρία Βέλα, αγαπητοί συνάδελφοι, αν θέλει να λάβει απόφαση ε, το Κοινοβούλιο για το πακέτο κινητικότητα σήμερα, ε, τότε θα διαρκέσει η αβεβαιότητα για το μεταφορικό τομέα. Ζητώ συγγνώμη. Ε, έχει πολύ θόρυβο στην αίθουσα. Δεν μπορώ να ακούσω καν τον εαυτό μου. Σας ευχαριστώ. Λίγη ησυχία λέει η Πρόεδρος. Παρακαλώ καθίστε ή αν θέλετε να συζητήσετε εκτός του ημικυκλίου. Σας παρακαλώ. Και για τον κύριο Μποβέ ισχύει αυτό. Κύριε Μποβέ. Η ε, κυρία Σόιντροβα, συνεχίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, επί Αυστριακής Προεδρίας ε, καταφέραμε να διαπραγματευτούμε συμβιβασμό στο Συμβούλιο για το πακέτο κινητικότητας. Και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι σε θέση να καταλήξει και αυτό σε παρόμοιο συμβιβασμό. Ξέρουμε ότι η οδηγία περί αποσπάσεως εργαζομένων προβλέπει ότι θα υπάρξουν νέοι κανόνες και συνθήκες που θα καθοριστούν για τους μεταφορείς και για τους οδηγούς φορτηγών. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα διοικητικής μορφής όσον αφορά τις παραβιάσεις των ε, κανόνων των συνθήκων. Χρειάζεται συμβιβασμός. Ο κ. Καπούτο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το πακέτο κινητικότητας πρέπει να εγκριθεί διότι δίνει ωφέλη και ανταγωνιστικότητα στον τομέα παραδείγματο χάρη στο cooling off για να αποφευθεί το καμποτάστο συστηματικό ε, όσον αφορά τι διεθνεί μεταφορέ και να έχουμε επίση και τον ΕΦΗ e ταχογράφο δεύτερη γενιά από το 2022. Όλα τα μέτρα που θα επιτρέψουν ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών στην Ευρώπη, εγγυούμενα όμω τα μέτρα την κοινωνική προστασία των εργαζομένων σε όλα τα κράτη-μέλη και θεμητό ανταγωνισμό. Η εναλλακτική είναι να βρεθούμε στο χάο με νομοθεσίε διαφορετικέ σε κάθε κράτο μέλο ε, και δεν θα είναι περισσότερη Ευρώπη και δεν θα είναι καν ενή αγορά. Όμω πιστεύω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία για το χρόνο οδήγηση και ανάπαυση για να υπάρχει μεγαλύτερη οδική ασφάλεια. Μία ανισόρροπη ε, κατανομή του χρόνου οδήγηση και ανάπαυση σημαίνει ότι οι συνθήκε θα έχουν άμεσε ε, συνέπειε για τι συνθήκε εργασία. Με περισσότερη κόπωση, λιγότερη συγκέντρωση, ε, μεγαλύτερη δυσκολία ανάκτηση των δυνάμεων και προβλήματα για του εργαζομένου και όλου του χρήστε των δρόμων. Λοιπόν, σας παρακαλώ και πάλι ησυχία. Παρακαλώ ησυχία. Και ε, ο κύριος Σόγκορ έχει το λόγο τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα με το πακέτο κινητικότητα δείχνει ότι δεν έχει καμία έννοια να συνεχίσει η εξέτασή του τώρα, ιδιαίτερα αν πρόκειται να το κάνουμε βεβαιασμένα. Κατά αυτή τη θητεία ήταν ε, από την αρχή στραβό το κλίμα. Αντί να κατηγορήσουμε και να τιμωρήσουμε ορισμένα εθνικά μέτρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέδειξε αυτή την περιοριστική πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρόταση αυτή δεν συμμορφούνται με βασικά κριτήρια για οποιοδήποτε νομοθέτημα. Πρώτα απ' όλα είναι κατά των αρχών της ε, ενιαίας αγοράς, πνίγει τον ανταγωνισμό, κάνει διακρίσεις ε, κατά μεγάλο αριθμό κρατών μερών, ε, πετάει στα σκουπίδια τα περιβαλλοντικά θέματα, με κανένα τρόπο δεν υπέρ των συμφερόντων των συμπολιτών και της Ένωσης. Ας κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε από λίγο πιο μακριά το θέμα, θα δούμε ότι ο προστατευτισμός θα μειώσει την ανταγωνιστικότητά μα. θα δημιουργήσει μονοπόλια, θα αυξήσει τις εκπομπές καυσαερίων και, θα, και τις τιμές για του καταναλωτές και θα διχάσουμε την Ευρώπη στα δύο. Οπωσδήποτε το πακέτο αυτό θα πρέπει να πάει στην επόμενη θητεία. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, ο κύριο Μπουσόη. Μπουσόη, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαιρετίζω την απόφαση του Πρέδρου Ταγιάννη να εφαρμοστεί το άρθρο 175 και να επαναπεμφθεί το πακέτο αυτό στην Επιτροπή. Κάνω έκκληση στη σοφροσύνη όλων των συναδέλφων, γιατί το πακέτο αυτό στην πραγματικότητα είναι δώρο για τους αντιπάλους της Ευρώπης. Οι οδικές μεταφορές, να μην το ξεχνάμε, είναι η κύρια πηγή εισοδήματο για δεκάδες ε, χιλιάδες οικογένειες εργαζομένων στις ε, περιφερειακές χώρες. Δεν είναι ισορροπημένη συμφωνία. Θα κατακαιρματιστεί η αγορά μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Πρέπει να υπάρξει επανεξισορρόπηση μεταξύ των καλών συνδικών εργασίας για τους οδηγούς, σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας, αλλά παράλληλα σεβασμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και των υπηρεσιών εντό της Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κράμπερ. Σας παρακαλώ να σέβεστε τον χρόνο σας. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Το ότι έχουμε τέτοια πίεση χρόνου είναι ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Γιούνκερ και ο Τίμερμανς για δύο χρόνια δεν επέτρεψαν στην Επίτροπο να υποβάλει τις προτάσεις αυτέ. Τότε θα είχαν περισσότερο χρόνο να τι συζητήσουμε αν είχε γίνει αυτό. Και φυσικά πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι. Αλλά έχουμε ταχυγράφου. Πριν από 15 χρόνους, χρόνια ήδη του είχαμε. Η Κομισιόν το 2036 ε, πρέπει να είναι υποχρεωτική η ταχυγράφη και ευτυχώ που είπαμε εμεί ότι πρέπει να είναι το 2024. Αυτοί οι νόμοι δεν λειτουργούν. Ξέρουμε ότι γίνονται πολλές απάτες και αυτό, επί, αυτό δημιουργεί κινδύνους για την οδική ασφάλεια και αν είναι δυνατόν πρέπει αυτοί οι ευφυείς ταχυγράφοι να αρχίσουν να ισχύουν από το 2022 και ολοκληρώνουμε τη διαδικασία Catch με τον κύριο Γκουόγκα. Ευχαριστώ πολύ να μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ χαμηλέ οι συντάξει ορισμένε χώρε. 300 ευρώ. Όλοι θα θέλαμε γερμανικού μισθού, αλλά δεν του έχουμε. Μην σκοτώσετε τι χώρε που είναι περισσότερο υπέρ τη Ευρώπη. Με αυτή την άθλια οδηγία, αθλιότατη, η οποία θα οδηγήσει τι ε, επιχειρήσει ε, σε πτώχευση και του ανθρώπου στην ανεργία. Θέλουμε καλύτερο επίπεδο μισθών, αλλά αυτό παίρνει χρόνο. Α εργαστούμε όλοι μαζί για να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη όπου όλοι να έχουμε καλέ αμοιβέ. Αλλά μην κλείσετε τι επιχειρήσει μα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, έτσι ολοκληρώνει τη διαδικασία Catch the Eye. Κύριε ε, Βέλα, σας παρακαλώ και εσείς να σεβαστείτε τον χρόνο σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές. εκ μέρους του Επιτρόπου Μπίλσο θέλω να σα ευχαριστήσω για τη σημερινή συζήτηση. Όλα τα στοιχεία των διαπραγματεύσεων βρίσκονται στο τραπέζι τώρα και ήρθε η στιγμή να ψηφίσουμε. Το πακέτο κινητικότητα θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα προσφέρει επίση ισότιμε συνθήκε για τι επιχειρήσει με ομοιόμορφου κανόνε και βελτίωση των συνθήκων εργασία για του οδηγού και επίση θα ενισχύσει και τι δυνατότητε για ελέγχου. Αντιμετωπίζει πολλά από τα γνωστά προβλήματα του κλάδου σήμερα. Και επιπλέον, τη απουσία ε, νέων ευρωπαϊκών κανόνων θα ε, οδηγηθούμε σε χειρότερες συνθήκες και με κοινωνικό ντάμπινγκ, με κατακαιρματισμό και προστατευτισμό όλο και περισσότερο. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Για κάποιες επιχειρήσεις το πακέτο θα προσφέρει σταθερές και προβλέψιμες συνθήκες και θα αποφύγει κανόνες ασυντόνιστους μεταξύ των χωρών μελών που πλήττουν την εσωτερική αγορά. Επίσης, το ποια έγγραφα θα πρέπει να ετοιμάζονται. Όλα αυτά θα είναι πιο σαφή και συγκεκριμένα κριτήρια και θα αποφύγουμε το φαινόμενο που όλο και αυξάνει τον επιχειρήσουμε εικονική έδρα. Όπως επίσης και τις πρακτικές συστημικού ε, εσωτερικού ενδομεταφορών μάλλον. Θα πρέπει επίση να είναι σαφέ και θα γίνει με αυτή τη ε, συμφωνία το ποιοι είναι οι κανόνε και ποια αντέγραφα που πρέπει να ετοιμάζονται. Επίση, θα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ψηφιακοί τρόποι υπέρ τη ασφάλεια και για την δήλωση τη απόσπαση. Για του οδηγού επίση το πακέτο προσφέρει ωφέλη, γιατί οι κανόνε απόσπαση θα εφαρμόζονται σε αυτού με κατώτατου μισθού και συγκεκριμένε συνθήκε στις χώρες που του φιλοξενούν. Επίσης, μετά από τέσσερις εβδομάδες θα μπορούν να επιστρέφουν σπίτι τους. Οι συνθήκες επίσης για τους ε, κανόνες εβδομαδιαίας ανάπαυσης και ότι οι εργοδότες πρέπει να πληρώνουν για την ανάπαυσή τους κάθε τόσο. Όλα αυτά θα βοηθήσουν να μην υπάρχει υπερβολική κόπωση των οδηγών, άρα είναι υπέρ της οδικής ασφάλειας. Επίσης, το μέτρο αυτό προσφέρει και περισσότερη ασφάλεια με τους ταχογράφους, με τον εντοπισμό τοποθεσίας και ενισχύεται και η διοικητική συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά έγγραφα για να ελέγχονται οι κανόνες δομεταφορών και για να διευκολύνονται ε, οι έλεγχοι της ασφάλειας. Ξέρουμε ότι πολλά από αυτά τα σημαντικά μέτρα ε, καταρχήν βρίσκουν σύμφωνους όλους τους ευρωβουλευτές, αλλά για τα άλλα ε, προτείνουμε να στηρίξετε τους συζητητές που πιστεύουμε ότι πετυχαίνουν μια καλή ισορροπία. Επίγει να διασφαλίσουμε ένα θετικό αποτέλεσμα όσον αφορά το πακέτο αυτό και αυτό πριν από τις ευρωεκλογέ. Η κατάσταση του κλείδου στην Ευρώπη, οι συνθήκε εργασία των οδηγών μα και το περιβάλλον μέσα στο οποίο δρούν οι επιχειρήσει μα είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα για να τα αφήσουμε σε ένα status quo για χρόνια που δεν ξέρουμε και πόσα θα είναι. Η κατάσταση είναι κρίσιμη και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ πολύ τους εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ευρωβουλευτές. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Κίλονεν, για να ολοκληρώσετε παρακαλώ. Έχετε το λόγο κύριε Κίλονεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Φτάνουμε στην τελική ευθεία του μαραθώνα. Φτάνουμε στον τερματισμό και ελπίζω το Προεδρείο να έχει το θάρρος να θέσει προς ψηφοφορία το πακέτο την επόμενη εβδομάδα στη Μήνη Ολομέλεια και να σταματήσει αυτή η κολυσιεργία. Ε, ανέφεραν οι συνάδελφοι ότι ήταν πολύ δύσκολο να αναγνωστούν αυτές οι τροπολογίες λόγω του αριθμού τους. Θέλω να πω ότι αυτές οι τροπολογίες κυκλοφορούσαν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη για περίπου δύο χρόνια. Τίποτα δεν άλλαξε σε σημαντικό βαθμό. Κάποιες ομάδες διαμαρτυρήθηκαν για το γεγονός ότι δεν τις επιτράπει να συμμετάσχουν επαρκώς. Να πω στο ENF ότι αν δεν συμμετέχετε σε καμία συνεδρίαση των σκιωδών το πρώτο εξάμεινο, πιστεύω ότι αυτό δείχνει ότι δεν είσαστε και υπερβολικά ενθουσιώδεις. Κάποιοι έχουν εδώ τις δικές τους κουβέντες και συζητήσεις. Θα ήθελα να πω ότι πρέπει να Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι πρέπει να συνεχίσουμε σωστή προσέγγιση. Και να πω και ένα τραγούδι. Κύριε Κάμπ θα μπορείτε να σταθείτε στο επίπεδο της προηγούμενης ομιλήτριας. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, Ναι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ξέρετε, πολλοί το λένε βέβαια, ε, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι η συζήτηση που είχαμε ήταν πάρα πολύ καλή. Και η συζήτηση αυτή έδειξε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το πακέτο κινητικότητας αριθμός 1 είναι διχασμένο. Και τώρα πρέπει να φροντίσουμε να μην πάρουμε τις κακές αποφάσεις στην κακή στιγμή. Και επειδή συνάδελφοι, Ερτούκο, Μιτσελίτσκα, Τελίσκα και ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι λένε, λένε ότι έχουμε συμβιβασμούς οι οποίοι δεν είναι που δεν ισχύουν, δεν είναι γεγονός. Υπάρχουν συμβιβασμοί για το καμποτάζ του Ισμαήλ Ερτούκ. Και τώρα, γιατί είμαστε σε δύσκολη κατάσταση εδώ, γιατί η Επιτροπή Μεταφορών, και εντάξει μπορεί να φταίω κι εγώ, δεν κατάφερε να πετύχει συμβιβασμούς, να τους εγκρίνει. Και αν συνεχίσουμε έτσι, είναι πάρα πολύ κακό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Και τέλος, ο κύριος Έρτουγκ. Ευχαριστώ, συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι η συζήτηση την τελευταία μία μισή ώρα απέδειξε άλλη μια φορά την αναγκαιότητα να υπάρξει μια λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σας διαβεβαιώ όλους όλους τους αδέλφους εδώ ότι τις επόμενες ε, μέρες θα τις αξιοποιήσω άλλη μια φορά για να επιδιώξω να υπάρξει λύση. Και καλώ όλους τους συναδέλφους να επιχειρήσουμε με ανοιχτό πνεύμα να συνοηθούμε με βάση τις προτάσεις που θα κάνω. Και επαναλαμβάνω, βρήκαμε σωστούς συμβιβασμού. Μπορεί να μην αποδεκτεί από όλους, αλλά θα ξαναπροσπαθήσουμε. Και ως εισηγητής και ως συντονιστής των σοσιαλιστών σας διαβεβαιώ ότι θα επιδιώξω να καταλήξω σε συμβιβασμούς. Αλλά στόχος μας πρέπει να είναι να εγγυηθούμε ότι θα ολοκληρωθεί και θα εγκριθεί η νομοθεσία πριν τη λήξη της θητείας, γιατί χρειαζόμαστε σωστή νομοθεσία για τους οδηγούς και ιδιαίτερα για τις έντιμες εταιρείε. Αυτό είναι το καθήκον μας και πρέπει να το κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Η κοινή συζήτηση έληξε και η ψηφοφορία θα γίνει στην επόμενη περίοδο Λομέλειας. Έχω μια ανακοίνωση. Ο κ. Γιάζεκ Σαριοσβόλσκι εγκαταλείπει τους μη γεγραμμένους βουλευτές και προσχωρά στην ομάδα ECR από τις 27 Μαρτίου του 2019. E Ξεκινάμε με τις ψηφοφόρειες. Έκθεση Μιχαήλοβα πόροι για το ειδικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Μία ψηφοφορία ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια. Η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου έτσι ολοκληρώνεται. Έκθεση Βέγκας και και αυτή η μοναδική ψηφοφορία ονομαστική που ξεκινάει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Έκθεση Μιχαήλοβα. Προϊόντα τα οποία δίνονται να τύχουν απ... απαλλαγής ή μείωση τη εισφοράς θαλάσση. Μοναδική ψηφοφορία ονομαστική που ξεκινάει. Τέλος. Εγκρίνεται. Έκθεση Πανζέρι Πρέντα Έγκερ Γκέρενς. Μηχανισμός γειτονίας ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας. 553 553-55-51. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε στην όμως... Λοιπόν, στην πρώτη ομάδα τροπολογιών, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 35 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 41, πρώτο τμήμα υπέρ, Θέλετε να κάνουμε μια, έναν έλεγχο, έναν έλεγχο για το δεύτερο τμήμα. Καλώς, ας το κάνουμε λοιπόν. Για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 35, ε, άρχεται η ψηφοφορία. La votazione è chiusa. Approvato. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 182 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 190 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 336 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 479 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 537 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 538 ονομαστική ψηφοφορία έρχεται. Πέρας. Α, απορρίπτεται. Τροπολογία 84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 539 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Α, απορρίπτεται. 540. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 541 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Ας κάνουμε έναν έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ο έλεγχος. Τέλος. Απορρίπτεται με μεγάλη διαφορά. Τροπολογία 109. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 542. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 543. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται. 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 544 ονομαστική κλίση ξεκινάει. Τέλος. Απορρίπτεται. 545 D. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 132-136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 546. Ονομαστική κλίση ξεκινάει. Πέρας. Απορρίπτεται. 279 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 547 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 359 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 548 D, ονομαστική κλίση, ξεκινάει. Πέρας. Απορρίπτεται. 415 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 549 D, ονομαστική κλίση που ξεκινάει. Πέρας. Απορρίπτεται. 454 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 550D. Ονομαστική κλίση ξεκινάει. Τέλος. Απορρίπτεται. 465 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 553 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 466 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 555 555 υπέρ συγγνώμη 555 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία Πέρασε. απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει. Τέλος. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού περιεχομένου 552 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 536 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 554 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος που ξεκινάει. Τέλος. Απορρίπτεται. Η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου ολοκληρώνεται λοιπόν. Συγχαρητήρια στους ε, εισηγητές. Και τώρα, τελευταία ψηφοφορία. Έκθεση Σαλαφράνκα Σάντσες Νέιρα Φλέκενστάιν. Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας. Ζήτησε το λόγο ο συνάδελφος Μακάλιστερ. Όχι. Εγώ λάθος κατάλαβα φαίνεται. Τροπολογία 130, ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει. Τέλος. Απορρίπτεται. Πάμε στο σχέδιο νομοθετικής πράξης. Πρώτη ομάδα ε, τροπολογιών υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία προφορική του συναδέλφου Σόλτες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Έχω προφορική τροπολογία. Ένα, δύο, τρία που αφορούν τα άρθρα 7, παράγραφος 5, γράμμα G. Να αντικαταστήσουμε τις λέξεις μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος με τις λέξεις αντιμετώπιση αλλαγής του κλίματος. Σύμφωνα το κουβεντιάσαμε και συμφωνήσαν οι δύο συνσηγητές. Ευχαριστώ κύριε Σόλτσες. Υπάρχει αντίρρηση όσον αφορά την προφορική τροπολογία του κυρίου Σόλτες. Όχι. Λοιπόν, ψηφίζουμε την τροπολογία 123 που τροποποιήθηκε όπως μας παρουσίασε και ο Σόλτες. Υπέρ παρακαλώ. Ε, κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει η τροπολογία 58, τροπολογία 124 υπέρ, παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 125 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 126 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 127 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 128 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει πέρας εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία συγχαρητήρια λοιπόν στους εισηγητές εμείς σταματάμε εδώ θα κάνουμε μια πάυση δύο λεπτών και μετά θα προχωρήσουμε στις επεξηγήσεις ψήφων. Ευχαριστώ.